υποδεχθώ εξ ονόματο όλων μας αρμενική αντιπροσωπεία που συμμετέχει στη 14η συνέλευση της κοινή ε, ε, συνέλευσης συνεργασίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αρμενίας. Καλώς ήρθατε. Κυρίως καλώς ήρθατε εσείς κύριε Φαρμανιάν που προεδρεύεται. Θα παρευρεθείτε σύντομα στη συνεδρίαση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ελπίζουμε η συνελευση τη κοινη συνέλευση συνεργασία ευρωπαικου κοινοβουλιου αρμενιας Καλώ ηρθατε Κυρίω καλώ ηρθατε εσεί, κυριε Φαρμανιά που προεδρεύετε. θα παρευρεθειτε συντομα στη συνεδριαση τη επιτροπη πρόσφατα και οι ανταλλαγέ απόψεων που θα έχουμε αυτέ τι μέρε να μα επιτρέψουν να πάμε πιο πέρα. Το θέμα που εξετάζουμε σήμερα είναι ο κατηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, αυτή την ημέρα της, που είναι η διεθνή ημέρα κατά τη μορφή αυτή βία. Καλώ ήρθατε λοιπόν και. Ο λόγο στην κυρία Κοράτσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επιτροπέ, φίλε.